Herzlichen Dank. Merci, λέει ο πρόεδρος. Ναι, με συγχωρείτε που άργησα, ήμουνα στην Χάγη, στην Κόζακ, για να συζητήσουμε το, τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το μεταναστευτικό και πρόσφυγες. Χτες συζητήσαμε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής. Για να μπορέσουν να συζητήσουν και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι αυτή η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη ψηφοφορία μας. Κοινή Ευρωπαϊκή Λίστα Ασφαλών Φόρων Προελεύσεως. Έχει ο κύριος Ράντος, ο εισηγητής, κάποια παρατήρηση. Όχι, ξεκινάμε τις φωτορίες. Δύο, τρία, τέσσερα. Υπέρ, κατά, αποχές απερίφθησαν. Εξήντα υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. ενα υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. No, but there are some from other groups. We cannot do that. Okay. Να κάνουμε όλες τις σαφοζέρ σε αμπλοκ. Κύριε Σαφοζέρ, συμφωνείτε. Υπέρ, παρακαλώ. Εκθέσει Σαφχάουζερ, παρακαλώ. Τροπολογία Σαφχάουζερ, υπέρ, κατά, αποχές. Καμία αποχή. Απερίφθη. Και τροπολογίες. 63 υπέρ κατά 23 υπέρ 30 κατά. 65 ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. 24 υπέρ 29 κατά 4 αποχές απερίφθη 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 74 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 83. 82 δύο 23 υπέρ, 33 κατά απερίφθη. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 77 υπέρ. Κατά. 78 συγγνώμη. 87 συγγνώμη. Απερίφθη. Μετά καταπίπτει, 85 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καστάλντο Χατζηγεωργίου Βαλέρο τώρα, χωρίς την ε, τροπολογία Σοφοζέχ, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. Συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η 10 καταπίπτει. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 17 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 όχι, την 23 επαληθεύουμε. 22 υπέρ 35 λέει ο μιλητής. Απερίφθη. 22 υπέρ κατά άποχες. Απερίφθη. 24 υπέρ κατά απεούχες. Απερίφθη. 25 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. 26 υπέρ, οι λοιπές ψήφοι 32. 26 κατά, υπέρ, κατά. Αποχές, επαληθεύουμε. 26. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, οι λοιπές 27. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. με σμάκερ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 ψήφι υπέρ, λέει ο ομιλητής. 11 κατά 18 αποχές. Συγχαρητήρια στον συγητή. Την συγγετρία. Και τώρα... Έκθεση Νόρικα Νικολάη. Παρατηρήσεις. Τη εισηγητρίας όχι. Μία η ψηφοφορία. ή δύο. τροπολογίε ένα και δύο. Κατά. Απερίφθησαν ψηφοφορία ηλεκτρονική τώρα για την ε, για το σύνολο. ψηφοφορία. 51 ψήφοι υπέρ. 5 ψήφοι κατά, 2 εποχές εγκρίνεται. Και τώρα η μερίσια διάταξη σημείο 15. Εδώ έχουμε τον Bruce Strokes. Έρευνα του Κέντρου Ερευνών Pew Research Center για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ. Μπρούς, έλα να κάτσεις. How are you in town?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 He will become my successor. Okay. Should I start or what do we yeah. do? You're grooming him. You're grooming him. I, I would like to thank you all for the... Να σας ευχαριστήσω όλους θα ήθελα πρώτα απ' όλα για την τιμή και την ε, μεγάλη αυτή ευκαιρία να σας παρουσιάσω μερικά από τα πιο πρόσφατα στοιχεία δια δημοσκοπήσεων που έχουμε διαλεργήσει για το πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τον κόσμο. Είναι παλιός φίλος ο πρόεδρος και εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του. Αυτή, η... αυτή είναι μια έρευνα που κάνουμε αντίστοιχη με αυτή που κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρωτούμε τους Αμερικάνους πώς βλέπουν τη θέση τους στον κόσμο. Και σωστά ήταν πολύ ενδιαφέρον να δουν οι Ευρωπαίοι πώς βλέπουν τη δική τους θέση στον κόσμο, ώστε να συγκρίνουμε και τις δύο αυτές αντιλήψεις ένθεν και εκείθεν του Ατλαντικού θα δώσουμε επίσης στοιχεία και για τους Ιαπωνέζους και τους Κινέζους, τη συνέχεια τους Ινδούς. Όλα αυτά γίνονται από το κέντρο έρευνας Πιού, που όπως ξέρετε είναι ένα κέντρο για δημοσκοπήσεις κοινή γνώμης που εδράζεται στην Washington. Δεν ε, έχουμε σαν στόχο <clears throat> το να υποστηρίξουμε κάποια άποψη. ανακαλύψαμε το ένα και ένα και ένα, αλλά δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε ότι το άθροισμα είναι τρία. Οι πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο των πολιτικών δημοσκοπήσεων γνωρίζουν για αυτά τα πράγματα που σας λέω. Πρώτη διαφάνεια. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να βρούμε το βαθμό ε, απομονωτικής στάσης, ε, προστατευτισμού πολυμέρειας ε, έναντι μονομέρειας, όλα αυτά τα λέμε για τους Αμερικανούς οι οποίοι ήταν ε, περισσότερο υπέρ της απομόνωσης και εμείς θέλουμε να πούμε ότι είμαστε σαν τους ε, Αμερικανούς, μας ενδιαφέρει το ελεύθερο εμπόριο. Όπως βλέπετε λοιπόν από αυτή τη διαφάνεια την οποία οι διερμηνείς βέβαια δεν βλέπουν και δεν έχουν στη διάθεσή τους η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και θεωρεί ότι και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν. Ορισμένοι μονάχα θεωρούν πρέπει να βοηθήσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς για να δει αν είναι κανείς απομονωτικός ή όχι. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ευρωπαϊκή άποψη για οποιοδήποτε θέμα. Υπάρχει μεγάλη πολυμορφία και διαφορετικότητα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάμεσος στην Ευρώπη είναι 56% λέει ο μιλητής. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι λένε εμείς θα αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα και οι άλλοι τα δικά τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αντίστοιχος δείκτης είναι 57%. Στον δείκτη αυτό απομονωτισμού ή εμείς πρώτοι από τους άλλους κατά κάποιο τρόπο, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση, να έχουν παρόμοια άποψη. Τα πράγματα βέβαια έχουν αλλάξει αρκετά στι ΗΠΑ στον τελευταίο καιρό, δεν έχουν αλλάξει στην ε, Ευρώπη. Τα στοιχεία μας για την Ευρώπη ξεκινάνε το 2010 μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση. Φυσικά από τότε τα άτομα είναι περισσότερο εστιασμένα στα εσωτερικά τους εθνικά θέματα. Και γιατί είχε κάνει έρευνα, θα μας πείτε, σε 10 μονάχα ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας πω, δεν είχαμε λεφτά. Αυτή είναι η απάντηση ειλικρινής. Διαλέξαμε τις χώρες που εκπροσωπούν το 82% της ευρωπαϊκής οικονομίας, 80% του πληθυσμού. Το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό. Αλλά νομίζουμε ότι είναι ένα δίκαιο δείγμα το οποίο είναι εκπροσωπευτικό της άποψης που επικρατεί στην Ευρώπη. Στην επόμενη αόρατη διαφάνεια σας ζητούμε να συγκρίνετε την πολυμέρεια με την μονομέρεια στις διεθνείς σχέσεις. Θα πρέπει η χώρα μας να ακολουθήσει το δικό της εθνικό συμφέρον στην εξωτερική πολιτική ανεξάρτητα από αυτά που λένε οι συμμαχοί μας ή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία μας ζητούν οι συμμαχοί μας όταν σχεδιάσουμε την εξωτερική μας πολιτική, όπως Βλέπετε, οι Έλληνε λένε δεν μα νοιάζει τι θέλουν οι συμμαχοί μας, ενώ δύο τρίτα των Γερμανών λένε πρέπει να λάβουμε υπόψη τις απόψει των συμμάχων μας όταν χαράσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Στις ΗΠΑ 51% είναι μονομερείς στην προσέγγιση τους. Μόνο 42% έχουν μια πολυμεριστική άποψη. Γι' αυτό είμαστε και πάλι πολύ κοντά στους Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε εσωστρεφείς και πιο μονομερείς στην σκέψη μας για την εξωτερική πολιτική. Επόμενη διαφάνεια. Θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη ιδέα του πώς θεωρούν η άποψη για το ρόλο που παίζει η χώρα, μας στο, η χώρα τους στον κόσμο και αν θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό ο ρόλος αυτός πριν από 10 χρόνια. Και πάλι μετά από αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, οι Έλληνες είναι σε κατάσταση κατατονική και τα δύο τρίτα τους λένε ότι κάνουμε, έχουμε λιγότερο ρόλο από ότι στο παρελθόν, ενώ έξι στους δέκα Γερμανούς λένε πιο σημαντικό είναι ο ρόλος μας στον κόσμο μετά τα τελευταία 10 χρόνια. Θα σας αφήσω να κρίνετε εσείς κατά πόσον είναι ακριβείς αυτές οι αντιλήψεις. 46% <clears throat> των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ παίζουν τώρα λιγότερο σημαντικό ρόλο στον κόσμο από ό,τι έκανε πριν από 10 χρόνια και αυτό εξηγεί αυτούς οι οποίοι έχουν σύνθηματα όπως το Τραμπ κάντε πάλι την Αμερική μεγάλη γιατί υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί που λένε ότι δεν είμαστε αυτό που ήμασταν στο παρελθόν. Μπορείτε να κρίνετε εσείς αν συμφωνείτε ή αν πιστεύετε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Η επόμενη διαφάνεια είναι ένα είδος αντίφασης, εκτός αν κάτσετε να τη σκεφτείτε. οι Ευρωπαίοι ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι κάνει στο παρελθόν και του ρωτήσαμε μήπως θα έπρεπε κατά την άποψή σα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Και λένε όλοι ναι. Η αντίφαση είναι ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επίκριση για τη διαχείριση κρίσεων από το προσφυγικό ως την Ουκρανία από τους πολίτες. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ακόμα κάποιος ιδεαλισμός, κάποιος ρομαντισμός πίστης στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλύτερη εξήγηση γι' αυτό είναι πριν από δύο χρόνια ζητήσαμε από του πολίτες να μας πούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπανε μα είναι γραφειοκρατική και τα αλλά τουλάχιστον μας φέρνει η ειρήνη και ευμάρεια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι πραγματικά σκέφτονται ότι υπάρχει ακόμα μια οραματιστική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλανε να παίξει περισσότερο ρόλο δεν τους αρέσει αυτό που κάνει σήμερα, είναι επικριτικοί, αλλά ακόμα συμμετέχουν σε αυτό το κοινό ιδανικό. Πάντως δεν έχουν ε, χάσει την ελπίδα τους στην Ευρώπη οι άνθρωποι. Κάτι το οποίο επηρεάζει τις διατλαντικές σχέσεις είναι η εντύπωση ότι οι Αμερικανοί είναι προστατευτικοί και κλειστοί, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ η έρευνά μας δείχνει ότι είναι περίπου το αντίθετο. Αν ρωτήσετε τους Ευρωπαίους αν θεωρείτε ότι είναι καλό για τη χώρα σας να συμμετέχει στην παγκόσμια οικονομία, 56% ε, λένε ναι, και ιδίω σε χώρες όπως η Ολλανδία, οι χώρες, η Γερμανία. Μόνο 44% των Αμερικανών όμω έχουν την ίδια άποψη ότι η συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία κάνει καλό στην Αμερική. 49% λένε κάνει κακό. Αυτά τα στερεότυπα λοιπόν για τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους δεν ισχύουν απόλυτα. Κάτι ακόμα που θα <clears throat> ψάχνουμε πάντα στις έρευνες αυτές που κάνουμε στην Ευρώπη είναι το κατά πόσον υπάρχουν περιφερειακές διαφορές. Και βλέπετε εδώ στην επόμενη διαφάνεια ότι υπάρχει συνεχής διαφορά στις απόψεις, κοινή γνώμη στην Γαλλία και στη Γερμανία εξακολουθεί οι Γερμανοί και οι Γάλλοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Κάτι ακόμα που είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ βορείων και ερωτήρων. Αλλά φαίνεται ότι οι Ισπανοί στην εκείνη τους ε, γνώμη μοιάζουν πολύ σαν τους ε, Βόρειο σαν τους Ολλανδούς, τους Σουηδούς, τους Γερμανούς, όχι σαν τους, σαν Ιταλούς και τους Έλληνες. Οι Ισπανοί από εσά ξέρουν καλύτερα πράγματα τη χώρα αυτή από μένα, αλλά αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα περάσω την επόμενη διαφάνεια, γιατί έχουμε ήδη μιλήσει για το πώ οι Ευρωπαϊκέ Αντιλήψει σχετίζονται και συγκρίνονται με τι Αμερικανικέ, αλλά ρωτήσαμε τον κόσμο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα σας. Αυτό που είδαμε είναι ότι το Ισλαμικό κράτος και η τρομοκρατία από το ISIS, το Ισλαμικό κράτος είναι το νούμερο ένα σε σχεδόν όλες τις χώρες. 80% των Αμερικανών λένε αυτό, ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή το Ισλαμικό κράτος. Κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μόνο 53% θεωρούν ότι είναι μεγάλη απειλή η κλιματική αλλαγή. αν πάτε στην επόμενη σελίδα και να δείτε θέματα τα οποία δεν ανησυχούν τον κόσμο. Λέμε για τις εντάσεις με τη Ρωσία. Μόνο οι Πολωνοί έχουν τέτοιους φόβους, η υπόλοιπη Ευρώπη δεν ανησυχεί τόσο πολύ. Η ανάδυση της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης, 29% μονάχα στην Ευρώπη θεωρούν ότι η Κίνα είναι μεγάλη απειλή. 50% των Αμερικανών θεωρούν ότι είναι κάτι τέτοιο. Σαν των Ισπανών <clears throat> και 43% ε, των Ελλήνων λένε οι Αμερικανοί είναι η κύρια απειλή για την Ευρώπη. Δεν ξέρω το πώς εξηγείται αυτό. Ο ευρωσκεπτικισμός είναι ένα σημαντικό θέμα. Ιδίως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση βρήκαμε για την άποψη της Ευρώπης μέσα στα τελευταία 15 χρόνια άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά υποστήριξης με την κρίση του ευρώ και κάπου μετά το 2012-2013 άρχισαν να ξαναανεβαίνουν και εφέτος είδαμε άλλη μία κάμψη σε σχέση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως υπάρχουν και άλλες απόψεις γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια πολύ απότομη πτώση σε πολλές χώρες. 17% στην Γαλλία, 16% στην Ισπανία. Αυτές είναι πολύ απότομες αλλαγές σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ βλέπετε το πόσο βλέπουν οι πολίτες θετικά ή αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, όπως βλέπετε, 22%, 27% των Ελλήνων υποστηρίζουν την Ευρώπη. Δεν είναι με εκπλήσει μετά από αυτά που έγιναν στην Ελλάδα, ενώ παρά το γεγονός ότι η πολωνική κυβέρνηση και η ουγγρική κυβέρνηση έχουν τις δικές τους διαφορές με τις Βρυξέλλες, το κοινό στην Πολωνία και την Ουγγαρία υποστηρίζει θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι νέοι έχουν πιο θετική άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι οι ηλικιωμένοι. Σε όλες τις χώρες <clears throat> και σε πολλές χώρες στατιστικά σημαντική αλλαγή, αλλαγή που φτάνει και στους 10 ποσοστιαίους πόντους. Αυτό δείχνει ότι οι νέοι δεν έχουν εγκαταλείψει την Ευρώπη παρά το υψηλό επίπεδο ανεργία σε πολλές από αυτές τις χώρες, ενώ είναι οι πιο ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν χάσει την πίστη τους στο ευρωπαϊκό όραμα. Επίσης, πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη ορισμένα θέματα, για να δούμε γιατί έχουν θετική ή αρνητική άποψη. Υπάρχει και πάλι μεγάλη ε, επίκριση σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπιση η Ευρώπη την ε, κρίση των προσφύγων, ιδίω από τις χώρες πρώτης γραμμής, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία <clears throat> και η Σουηδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι η, πρώτη, η χώρα πρώτης γραμμής γιατί έχουν πάρει πολλούς πρόσφυγες. Και έχουν θυμώσει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το λόγο. Τώρα έχουμε την ερώτηση για το πώς θεωρούν ότι χειρίζεται τα οικονομικά η Ένωση και αυτό το έχουμε ξαναρωτήσει στο παρελθόν. Συνεχίζονται οι επικρίσεις, ε, φυσικά οι πιο επικριτικοί είναι οι Έλληνες και οι Γερμανοί οι λιγότερο επικριτικοί. Δεν είναι φυσικό και αυτό, δεν εκπλήσει. Ε, οπότε έχουμε ε, αυτές τις επικρίσεις για την οικονομία αλλά και για την Ρωσία. Πώς χειρίζεται τις σχέσεις με την Ρωσία. Οπότε εδώ βλέπετε ότι οι απαντώντες απαντούν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς λόγους. Σε λίγο θα σας δείξω μια διαφάνεια όπου εμφαίνεται ότι έχουμε 69% των Ελλήνων που επικρίνουν τις ε, σχέσεις με τη Ρωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς τις χειρίζεται η Ένωση. Ε, αυτό όμως σημαίνει ότι είναι πολύ ενδοτική, πολύ αυστηρή. ιδέα δε ιδέα λένε ότι δεν τα πάει καλά με τη σχέση με τη Ρωσία ε, για τον ένα για τον άλλο λόγο αλλά στην άλλη διαφάνεια όπως θα δείτε μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση διότι εδώ ρωτήσαμε τους Ευρωπαίους θέλετε να είμαστε σκληρότεροι με την Ρωσία να έχουμε καλύτερες οικονομικές σχέσεις οι Σουηδοί είπανε όχι να είμαστε σκληροί με την Ρωσία να γιατί επικρίνουν την Ένωση δεν είναι αρκετά σκληροί και είπαν καλύτερες οικονομικές σχέσεις οι Έλληνε. <clears throat> Να γιατί επέκριναν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ αυστηροί με τους Ρώσους και εσείς με στην πολιτική του ζωή σας και ξέρετε ότι τα ανάμεικτα μηνύματα από τον κόσμο δεν είναι κάτι το εκπληκτικό. Απλώς εσείς πρέπει να τα ερμηνεύσετε και είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι Τώρα έχουμε το ερώτημα που ρώτησαμε όλους τους Ευρωπαίους γιατί θέλαμε να δούμε ακριβώς σε σχέση με το Brexit πώς αισθάνεται ο κόσμος. Δεν ρωτήσαμε τι θα ψηφίσετε τους ε, Βρετανούς γιατί θεωρήσαμε ότι το θέμα εδώ είναι αν θέλει κανείς περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη πιο αποκεντρωμένοι ή πιο κεντροκατευθυνόμενοι. Λιγότερη περισσότερη δύναμη στις πρωτεύουσες. Βλέπετε εδώ ότι δεν θα σας εκπλήξει ότι 65% των Βρετανών είπαν ότι θέλουν να ξαναγυρίσουν οι εξουσίες στο Λονδίνο. Γι' αυτό γίνεται και άλλωστε και το δημοψήφισμα. Αλλά μου φάνηκε ενδιαφέρον το ότι η μεγάλη πλειοψηφία σε πολλές χώρες λένε και εμείς θα θέλαμε περισσότερες εξουσίες να ξαναγυρίσουν στην πρωτεύουσά μας. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσουν στις 23 του μηνός οι Βρετανοί, η προβληματική θα συνεχιστεί στην Ευρώπη. Από τη μια μεριά περισσότερη ή από την άλλη λιγότερη Ευρώπη. Κάτι το οποίο θα πάει, ε, θα συνεχιστεί. Βλέπουμε εδώ πέρα η ε, αυστηρή, η ε, λιγότερο αυστηρή πολιτική. Ε, εδώ λέμε, ας πούμε, εάν βελτιωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, αυτό θα πρέπει να είναι άξονας της εξωτερικής μας πολιτικής ή όχι. Όπως βλέπετε, οι Ευρωπαίοι διαφωνούν από αυτού. Οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Ισπανοί θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα τα δικαιώματα. Δεν συμφωνούν οι Ούγγροι ή οι Πολωνοί με τούτο όμως και μέσα όρος είναι 42%. Περισσότεροι λένε ότι θα πρέπει να 42% λένε θα πρέπει να άξουν συγκεκριμένη πολιτική, 44% στις ΙΠΑ τώρα όσον αφορά τις σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τρία ερωτήματα. Τι γίνεται με τις επενδύσεις των εταιριών, τι γίνεται με τις περισσότερες εισαγωγές από αυτές τις χώρες και πώς βλέπετε την αύξηση της ξένης βοήθειας σε αυτές τις χώρες. 53% ήταν ο μέσος όρος. 83% κυμαίνεται που θέλουν οι Ισπανοί και 28% λέει η Ελλάδα για την αύξηση της ε, εξωτερικής βοήθειας. 48% είπε η Αμερική. Επομένως, βλέπουμε ότι λίγο περισσότερο από τους Αμερικανούς, οι Ευρωπαίοι θέλουν να αυξηθεί η ξένη βοήθεια. Ας είστε εσείς πιο κοντά στους στόχους του όσα ερμηνεύστε το. Για το ΝΑΤΟ επίσης. Υπέρ κατά. Αυτό το ρωτάμε κάθε χρόνο, άλλαξε τα τελευταία χρόνια και ο μέσος όρος λέει ότι είναι περισσότερο από τους Αμερικανούς υπέρ. 53 και 59% αντίστοιχα. Και εδώ όμως βέβαια υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις. 21% του κόσμου στις είπα, είπαν ότι δεν έχουν άποψη. Και έτσι που το στέλνει Department να κάνουμε κάτι, να ενεργήσουμε διπλωματικά μέσω του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι το ΝΑΤΟ άλλαξαν τα πράγματα με αυτή τη γενιά. Εγώ μεγάλωσα στον ψυχρό πόλεμο. Όλοι στο μυαλό του είχαν το ΝΑΤΟ. Και μετά την πτώση του τείχους έχουμε φρέσκες γενιές. Οπότε μειώθηκε και η σημασία του ΝΑΤΟ. Επίσης ένα από τα θέματα που αποτελούν συνεχή προβληματική σε Ευρώπη και Αμερική είναι οι αμυντικές δαπάνες. Βεβαίω εμεί ε, ποσοστία δίνουμε περισσότερα από τους Ευρωπαίους, σαν του ΑΕΠ. Βλέπετε όμως ότι οι Πολωνοί και οι Ολλανδοί θέλουν αύξηση. Οι Ιταλοί, Έλληνες, Ισπανοί δεν θέλουν αύξηση. Μεσο όρο είναι 33% για την αύξηση αμυντικών δαπανών. 35% το αντίστοιχο ποσοστό στη ΣΥΠΑ. Αφενός, αυτό δεν είναι πολύ υψηλό. Ποιο θέλει να οι νομικέ δαπάνε από την άλλη, όμω επί χρόνια ρωτάμε το ίδιο. Και το 35% στη ΣΥΠΑ είναι ιστορικό ρεκόρ για την περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τους δύο πύργους. Και υπήρχε και μια μηνότητα που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει αύξηση περισσότερο ρεπουμπλικάνοι παρά δημοκράτες. Είπαν ναι στην αύξηση. Επίσης, μεγαλύτερη απειλή θεωρήθηκε η τρομοκρατία. Η ερώτηση, να χρησιμοποιήσουμε το στρατό κατά της τρομοκρατίας. Είναι καλό ή θα ε, φουντώσει η τρομοκρατία να το κάνουμε αυτό. Όπως βλέπετε, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί πιστεύουν κατηγορηματικά ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο στρατός κατά της τρομοκρατίας και θα οδηγήσει αυτό όμως σε φούντομα της τρομοκρατίας. Και οι Ιταλοί, οι Ούγγροι ας πούμε λένε ότι δεν θεωρούν ότι η χρήση του στρατού θα φέρει αυτό λοιπόν και θέλουν χρήση του στρατού. Ε, εμείς, σαν κομπόδες, είμαστε διχασμένοι, 47% λένε ότι να χρησιμοποιηθεί ο στρατός κατά της τρομοκρατίας, 47% λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει περισσότερους τρομοκράτες. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι είμαστε διχασμένοι και αν ακόμα. Τίνουν οι Ρεπουμπλικάνοι να πούνε να χρησιμοποιούν το στρατό, οι Δημοκράτες λένε ότι όχι, έτσι θα έχουμε περισσότερους τρομοκράτες. Τα ξέρετε, τι να σας πω. Κάθε μέρα τα ακούτε από τους ψηφοφόρους σας γιατί θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά ή όχι. Και εδώ πέρα υπάρχει διχογνωμία αριστεράς και δεξιάς. Αν δούμε το φάσμα, οι δεξιοί τείνουν να πούνε ότι ας ασχοληθούμε με τα εσωτερικά. Οι αριστεροί τείνουν να πούνε ότι όχι, θα πρέπει να βοηθήσουμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται εκτός της χώρας. Και υπάρχει η ίδια διχογνωμία και όσον αφορά το ερώτημα περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Ως επιτοπλίστων, οι δεξιοί θέλουν οι εξουσίες να επιστρέψουν στις εθνικές κυβερνήσεις. Το θέλουν περισσότερο από τους αριστερούς. Όμως είναι το ανάποδο σε Ισπανία και Ελλάδα. Οι αριστεροί θέλουν περισσότερες αρμοδιότητες για την εθνική κυβέρνηση. Και αν δείτε την ανάλυση ανακόμα, βλέπετε ότι εδώ με ποιον ταυτίζονται σαν, σαν κόμμα, αλλά εγώ που δεν είμαι Ευρωπαίος, βλέπω ενδιαφέρον το τι γίνεται με τους οπαδούς του εθνικού μετόπου στην Γαλλία. Αυτή Εκεί, ζητούν περισσότερο οι σοσιαλιστές, περισσότερες αρμοδιότητες. Στην Πολωνία τώρα, 48% θέλουν το ίδιο να γυρίσουν εξουσίες στην Βαρσοβία και μόλις 19% της πλατφόρμας των ε, πολιτών. Και αυτά σε κάποια χώρα που υπάρχει πολύ σφιλό ευρωπαϊσμός. Θα πείτε αντίφαση. Ε, ναι, αλλά να, από προκύπτει το ενδιαφέρον από τα μηνύματα του κόσμου. Τώρα για το προσφυγικό. Ρωτήσαμε αν ακόμα. Κοιτάξτε τις απαντήσεις. Όπως λέτε, εδώ. Το εθνικό μέτωπο ανησυχεί περισσότερο από ότι το σοσιαλιστικό κόμμα για τους ε, πρόσφυγες. Το Φορτσά Ιταλία επίσης ανησυχεί περισσότερο από ότι το πιντή στην Ιταλία. Και βλέπετε στην τελευταία διαφάνεια ότι το Ποδέμος θέλει περισσότερο από τα άλλα κόμματα να επιστρέψουν η εξουσίες στην Μαδρίτη. Οπότε αν το δείτε ανακόμα θα καταλάβετε πώς διαμορφώνονται αυτά τα ζητήματα ανακόμα στην πολιτική. Αυτή η έρευνα σήμερα δημοσιοποιήθηκε και τον επόμενο μήνα θα έχουμε μία έρευνα για μουσουλμάνους, ε, Εβραίους, ε, ε, πρόσφυγες, εθνική ταυτότητα. Πώς θα είναι το κόσμο στην Ευρώπη για αυτό, τι πιστεύει, να είστε έτοιμοι. Και επίσης που συγκρίνεται τα σχετικά στοιχεία της Ευρώπης με τα Αμερικανικά και αντιστρόφως. Να είστε έτοιμοι για αυτή την έρευνα επομένως και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι όντως πολύ ε, ενημερωτική η έρευνά σας. Γνωρίζετε φαντάζομαι. Και ξέρετε ότι έχουμε μεγάλες τάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε και οι ηγέτες μας θα πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη ώστε να αρχίσει η εκπαίδευση των πολιτών να μην στηρίζονται μόνο σε αυτό που πιστεύουν οι πολίτες. Ιδάλλως θα φτάσουμε σε μια μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Κύριε Γκόμες, κυρία Φωτίκα, ευχαριστώ πολύ Μπρούς. Πολύ ενδιαφέροντα για μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κυρία Μέλκα τα δώσατε αυτά. Στην κυρία Μέρκελ. Γιατί έχει δείξει η έρευνα ότι, όπως καταγράφεται, η πιο ισχυρή ηγετική στάση της Γερμανίας δεν έχει οδηγήσει σε καλύτερη ηγετική θέση και ηγεσία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβει υπόψη. Οι πολίτες διατηρούν την, ε, τις προσδοκίες τους. Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου φαντάζομαι η Πορτογαλία θα έχει απαντήσει αντίστοιχε με αυτέ της Ισπανία εκτό από το ότι θα ήμασταν λιγότερο κατά των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Είναι ενδιαφέρον όμω ότι οι Ισπανοί και οι Γερμανοί έχουν υψηλότερα ποσοστά πολιτών που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια ισχυρή δύναμη και να ε, επιδιώκει ένα καλύτερο κόσμο. Αυτά πρέπει να τα δει η κυρία Μέρκελ. Πρέπει από τα λάθη μας να δασκόμαστε. Και όλοι μας έχουμε διαπράξει σφάλματα. Τα χειρότερα μάλιστα είναι αυτά στην οικονομία. Αλλά ας κοιτάξουμε τι προσδοκίες τρέφουν οι πολίτες. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο για δουλειά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ενδιαφέρον το ότι χώρες όπου κάποιες δυνάμεις χρησιμοποιούν ως εργαλείο προπαγάνδας στους πρόσφυγες βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές, παρότι δεν υπάρχει πραγματική απειλή, ανταποκρίνονται στην απειλή. Η Πολωνία έχει ωφεληθεί από την οικονομική κατάσταση. Έχει όμως έντονα συναισθήματα για την Πολωνία και θεωρεί, για την Ρωσία και θεωρούν οι Πολωνοί ότι δεν τους παρακολουθούν οι λοιποί. Αλλά ταυτόχρονα έχουν και μεγάλες ανησυχίε για το προσφυγικό και ότι η Πολωνία δεν είναι από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την εισρωή μεταναστών ή προσφύγων. Από την άλλη χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή της υποδοχής προσφύγων δείχνουν μια πολύ πιο δεκτική και πεφωτισμένη θα έλεγα προσέγγιση των προσφύγων. Σας ευχαριστώ. Φωτσίκα. Ε, ευχαριστώ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση, ε, μια και με Πολωνή. Θα ήθελα να δώσω πληροφορία στην κυρία Γκόμες για το όσα είπα. Η Eurostat λέει ότι το 2014, αν δεν κάνω λάθος στα στοιχεία μου, η Πολωνία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η χώρα που απεδέχθη το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, λέει η ομιλήτρια από την Ουκρανία επί το πλήστον. Αλλά ναι, έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά. Κυρία Γκόμες, δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Φωτσίγκα, όχι, όχι, του αντίον, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει. Ανοχή ήταν το ζήτημα. Ε, εν εντάξει. Δεν δίνω συνέχεια. Ενημέρωση θέλω μόνο και μουσουλμάνους από την Τσετσενία. Δύο κύματα. Μένα ενδιαφέρον με ενδιαφέρει η αντίληψη η σχετική με τις αμυντικές δαπάνες. Αναχώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δυναμική της ε, θεώρησης αυτής είναι ανωδικές στάσεις ή όχι. Αναφέρατε τις ΗΠΑ και τις συνθήκες που επικράτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά στην Ευρώπη τι βλέπουμε. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε δεδομένα που να μιλούν για βούληση αύξηση των αμυντικών δαπανών. Μόνο στιγμιότυπο μπορώ να σας δώσω και όχι τάσεις. Ωστόσο πέρσι μια μελέτη μας ρωτούσε με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, εάν δηλαδή θα δέχονταν ο κόσμος να προσφέρει την αλληλεγγύη των ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από το ΝΑΤΟ. Δύο πράγματα έχω να απαντήσω. Πρώτον, ότι κανείς δεν είχε θέσει το ερώτημα πριν. Πράγμα το οποίο δείχνει μια ανευθυνότητα από τους υπεύθυνου. Γιατί δεν θέλω να ακούσουν σωστή απάντηση, γι' αυτό δεν έδωσαν την ερώτηση αλλά πάντως 56% των Γερμανών είπαν ότι δεν θέλουν ε, να αναλάβουν δράση δύναμη του άρθρου 5. Οι Γάλλοι μάλλον όχι, οι Ιταλοί μάλλον όχι, οι Βρετανοί μάλλον ναι, οι Αμερικανοί μάλλον ναι, σε μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα η συμμαχική δομή και η εντύπωση που έχουμε για αυτήν φαίνεται να δίνει κάποια αποτελέσματα. Ακόμη και μόνο με την επίκληση του άρθρου 5 ο πολίτης, όχι ίσω η ελίτ, έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη και διαφορετική από τη ελίτ του για το τι σημαίνει αυτό το άρθρο. Και εκεί βέβαια φαντάζομαι ότι εστιάζεται και το εάν είναι διτεθειμένο ο πολίτης να διαθέσει δαπάνε για την άμυνα. Ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει τόσο μεγάλη υποστήριξη. Και αυτά κατόπιν των ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία. Όχι δηλαδή σε μια ανύποπτη στιγμή που θα λέει κανείς τι να το κάνουμε τον άτο. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω πως οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι τα προσφυγικά ρεύματα από την Συρία και το Ιράκ είναι μεγάλη απειλή για τις ΗΠΑ, ενώ έχουμε υποδεχθεί μέχρι 3.000 πρόσφυγες στο πολύ. Γελώ μεν, αλλά θα πρέπει να κλαίγω. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρώτο Πάσκου, είναι αδύρυτο και είναι στοιχείο κοινή λογική ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αντίληψη κινδύνου που οδηγεί σε περισσότερες αμυντικές δαπάνες. Φαίνεται να συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Είναι λιγότερο έντονο στη δική Ευρώπη όπου υπάρχουν πιο απομακρυσμένες απειλές. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι το έγγραφο αυτό θα σας διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Γιατί έχει γίνει μόλις τώρα δημόσιο από τον ομιλητή. Θα πάρετε λοιπόν αυτή τη μελέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ο κύριος Ντεφ Σούμπελ, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, για να μας παρουσιάσει την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Yes, a very good afternoon. Είναι εδώ, ναι, βεβαίως. Θέλετε να έρθω στο Πόντιο. Αν θέλετε, βεβαίω. Εντάξει, μπορείτε να μιλήσετε από εκεί όπω θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που μπορώ να αναφερθώ σήμερα για ένα θέμα που δεν έχει σταθεί πάντα εύκολο ζήτημα τα τελευταία δύο χρόνια για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερμπαϊτζάν. τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα στις σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Αζερβαϊτζάν, όπω ξέρουν όλοι οι δημονε για τη σχέση μα. Υπήρξε πραγματική καταστολή στην κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επικρίνει αυτή την καταστολή και αυτό οδήγησε σε αναστολή από το Αζερβαϊτζάν όλων των συναντήσεων που έλκονται από τη Συμφωνία σταθεροποίηση και συνεργασία και επίσης στις ε, πολυμερείς ε, συναντήσεις της ε, Ανατολικής γειτονία. Και ξέρετε ότι το Αζερβαϊτζάν έχει αποσυρθεί και από τις παρουσίες του στις συναντήσεις της Euronest. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσπάθησαν να κρατήσουν κάποιους διάβλους επικοινωνία ανοιχτούς. Ο κ. Ναμπρινίδης, ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πήγε στον Πακού το Φεβρουάριο, συνάντησε και κάποιους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν στη φυλακή, βέβαια εκείνη την εποχή. Ο Επίτροπος Χάν πήγε τον Απρίλιο στον Πακού πέρσι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. πήγε τον Ιούλιο πέρσι. Σε όλες αυτές τις επισκέψει εκφράστηκαν οι ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν, στο πιο υψηλό επίπεδο, προ τον πρόεδρο Αλίγεφ. Του τελευταίου μήνε όμω οι σχέσει μεταξύ των δύο μερών είναι κάπω πιο θετικέ και αυτό επιβεβαιώθηκε από την επίσκεψη τη ΥΠΑ, του, ΥΠΑ της εκπροσώπου στο Μπακού στις 29 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου. Και αυτό ακολουθήθηκε από κάποιες απελευθερώσεις των ε, ακτιβιστών υψηλού προφίλ, ακόμα και την άδεια να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ε, Γιούνους, ε, Λέιλα και Άριφ και ο Ίντιγκαμ Αλίεφ. Επανέρχομαι στις διμερείς μας σχέσεις. Στην ε, διάσκεψη της Ρήγας, τη διμερή συνάντηση κορυφής στη Ρήγα, το Αζερβαϊτζάν έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόταση για στρατηγική εταιρική σχέση που ουσιαστικά είναι τροποποίηση της τωρινής μας νομικής βάσης που είναι μια συμφωνία συνεργασίας και εταιρική σχέσης. Μετά από κάποια διαρευνητική επίσκεψη στον Πακού με επικεφαλής τον Τόμας Μάιες Χάτινγκ από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το Δεκέμβριο του 2015, όπου και οι δύο πλευρές προσπάθησαν να καταγράψουν το, την εμβέλεια και τις φιλοδοξίες της συμφωνίας που πρέπει να συναφθεί. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια νέα εντολή, η οποία θα δοθεί στο, από το Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι νέες διαπραγματεύσεις. Θα είναι φιλόδοξες αυτές οι νέε διαπραγματεύσεις, θα έχουν στεναρές ρήτρες για την κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και επίσης θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ κατάλογο δυνητικών χώρων συνεργασίας αμοιβαίου συμφέροντος. Αυτή η νέα συμφωνία μπορεί να είναι και μια λιδία λίθος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας γιατί θα δράζεται στην αρχή της διαφοροποίησης και θα επιτρέπει να είναι ορισμένες λύσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες σε κάθε χώρα χωρίς να θίγονται οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τονίστηκαν από την ύπατη εκπρόσωπο στην αρχή του χρόνου στην επίσκεψη στον Πακού, συναντήθηκε με τον προ... Πρόεδρο Αλίγη, από τον κύριο Μαμαριά, τον Υπουργό Εξωτερικών και μέλη και μέλη τη κοινωνία των πολιτών. Ήταν μεγάλη επιτυχία αυτή η επίσκεψη, διότι επανέφερε ένα επίπεδο εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και έχουν γίνει τώρα θετικά βήματα από το Αζερβαϊτζάν έκτοτε. Σε επίπεδο διμέρες το Αζερβαϊτζάν αποφάσισε να επανέλθει σε όλες τις συναντήσεις στα πλαίσια τη Συμφωνίας Εταιρικής και συνεργασία. Θα ξεκινήσουμε με τη συνάντηση Επιτροπή για το εμπόριο την ενέργεια και επίσης επιτροπές για τη δικαιοσύνη, για το διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επαφή ανθρώπων με ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν στον Πακού. Και το Αζερβαϊτζάν συμμετέχει σε όλες τις δομές της ε, πολυμερούς πτυχής της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Στις 3 Ιουνίου ήταν και η κοδεσπότη σε μια τέτοια συνάντηση. Η φιλοδοξία μας για αυτή τη νέα συμφωνία είναι η ενημέρωση της τωρινής μας νομικής βάσης και να αντικαταστήσει την προηγούμενη συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας, θα διευρύνει τη συνεργασία μας και σε νέους τομείς όπως είναι η πολιτική αεροπορία, η ψηφιακή οικονομία και συνεργασία στις ε, συνδέσεις μεταφορικού χαρακτήρα. Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε την επανάληψη της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από την επίσκεψη του, της κυρίας Χάουτουρο και του κυρίου Ντελίζε στο Μπακού, που είναι οι πρόεδροι της Αρτιστικής Επιτροπής και της πρόθεσης να υπάρξει συνάντηση Επιτροπής Συνεργασίας τον Σεπτέμβριο. Έτσι αυτό μπορεί να μας βγάλει από την κατάσταση στην οποία είμαστε υπήρξε και η θέληση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη συμμετοχή του Αζερβαϊτζάν σε ευρωπαϊκού φορεί και ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά είναι θετικά μηνύματα. Όλα αυτά έχουν εγκριθεί σήμερα, αν δεν κάνω λάθο, από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και αυτό είναι ένα πολύ θετικό ε, βήμα και πρέπει να σα πω πρέπει να σα εκφράσω την ικανοποίησή μου. επίση, 17 Μαρτίου, ο πρόεδρος έδωσε χάρη σε 48 κρατουμένους μεταξύ των οποίων 14 ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φασούλ Τζαφάροφ, ο Τόπιο Γιακούμποφ και ο Άννα Αρμαβάλη. Οι υποόρους απελευθέρωση του Ιντερ Καμαλή, του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που του να πάει στο Στρασβούργο, ήταν και αυτό θετικό. Και επίση το ζευγάρι Γιούνου που μπόρεσε να πάνε στο εξωτερικό και να έχουν ιατρική περιθέρψη και ξέρουμε ότι και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάστηκαν ιδιαίτερα για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Τελευταίο θετικό στοιχείο, η περίπτωση της Κατήγια Ισμαήλωβα, η οποία υπό όρους απελευθερώθηκε. Υπάρχουν κάποιοι ακτιβιστές των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί ξανά άνοιξαν και ήρθε η απαγόρευση ταξιδιού στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι δεν έχουν απελευθερωθεί όλοι οι κρατούμενοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Τι μπορούμε να δούμε λοιπόν ως αίτια αυτής της προσέγγισης. Προφανώς έχει να κάνει και με την εσωτερική κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν και ίσως και την οικονομική κατάσταση πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί πολύ, πολύ η ενεργειακά κυριαρχούμενη οικονομία του Αζερβαϊτζάν. Υπήρξαν δύο ε, υποτιμήσεις το 2015 του Αζερβαϊτζανικού Μανάτ. Έχει αυξηθεί η ανεργία αλλά και, η, και ο πληθωρισμός. Η άρση των κυρώσεων προς το Ιράν επίσης ξανήξαν ε, δυνατότητες και για το Αζερβαϊτζάν που είναι γείτονες και αυξήθηκαν όμως οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας κατά κάποιο τρόπο τούτο έκανε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Αζερβαϊτζάν πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτά οι θετικέ νότα τώρα και άλλα προβλήματα απομένουν και για των πολιτών, ε, τι γίνεται με τους ακτιβιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων, ακόμη κάποιοι αυτούς είναι στη φυλακή, τον Μάμαντοφ να αναφέρω ενδεικτικά έχει υπέρ του μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 έκτου το Συμβούλιο α, της Ευρώπης αποφάσισε να είναι πάγιο σημείο στην εμέσια διάταξη ε, ούτω ώστε να ασκηθεί πίεση στις αρχέ τη χώρα για να τον ε, ε, απελευθερώσουν και ο Γενικό Γραμματέα. Αποφάσισε να επικαλεστεί το άρθρο 52 για πρώτη φορά για την υπόθεση του τόσο ώστε να υπάρξει διερεύνηση. Υπάρχει και άλλη μία ε, ε, περίπτωση που αφορά κάποια διαδικασία γραφειοκρατική. Ε, σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία δεν μπορούν να ενισχύσουν τη χώρα οι δωρητές και είπε ότι εκπρόσωπο έθισε το πρόβλημα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο όταν έκανε αυτή την υψηλού επέδου συνάντηση. Η υπηρεσία εξωτερική δράση και η επιτροπή θα εξασφαλίσουν το ότι θα υπάρξουν καλύτερε συνθήκε, αλλά βέβαια θα πρέπει να βρεθεί μια ε, λύση ad hoc από την αντιπροσωπεία μα στο Μπακού. Οπότε εργαζόμαστε εντατικά στη συνεργασία με τι αρχέ χώρα. Βέβαια είναι και πολύ σημαντική η προστριβή στον Αγκόνο Καραμπάχ. Τον Απρίλιο εντάθηκαν οι εχθροπραξίες και διαπιστώσαμε ότι είναι δυνατόν αυτές οι προστριβές να γίνουν ε, εμπόλεμη ε, αναμέτρηση. Οπότε ξεκινήσανε κάποιες ε, διαπραγματεύσεις για να υπάρξει κάποια ρύθμιση και την Βιέννη 16 Πέμπτου σαντίθηκαν οι επικεφαλείς των κρατών και πήγε και η κυρία Σμιτ και στις 31 ε, Πέμπτου συνάντησε εκπροσώπους της ομάδας του Μίνσκ. Έγινε ε, με τους συμπροέδρους η κατάβαυση του πύρος ε, και βοήθησε και ο κύριος Ζάλμπα. Εμείς θα προσπαθήσουμε περισσότερο με τους συμπροέδρους, με την ομάδα του Μίνσκ, ούτως ώστε η Ρευτική Συμφωνία να υλοποιηθεί. Πάντως εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ειρήνευση και προσπαθούμε να ε, έχουμε μια εταιρική σχέση που θα βοηθήσει για να υπάρξει μίληση για τον αργόνο Καραμπάχ αυτό ε, θα ενταθεί σαν προσπάθεια όλο ένα και περισσότερο όσο εντείνεται η σύγκρουση. Είχαμε πάντως στις ε, στις διμερείς σχέσεις ένταση. Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξυπηρεθούν τα συμφέροντά μας και επίσης θέλουμε να αποφυλακιστούν η Ισμαήλωβα, ο Καντιέφ και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμα αλλά θεωρούμε ότι η κατάσταση όπως είναι σήμερα αποτελεί μια ευκαιρία για τις σχέσεις μας με το Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Η νέα συμφωνία είναι μια ευκαιρία να δοθεί μια όθηση στις επαφέ με τη χώρα και μια ευκαιρία να συζητήσουμε αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κρίσιμη στιγμή επομένω και η διπλωματία μας προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας, αλλά έχει σημασία να είμαστε συνεπείς και να ακούγεται η ενιαία η φωνή της Ένωσης. Είναι σημαντικό επομένω να υπάρχει συντονισμό στο τι μηνύματα στέλνουμε. Σε όσο γίνεται περισσότερη επίπεδα να δράσουμε, να ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδει ελευθερίε, οπότε θα πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τι αρχέ τη χώρα. Θα να προσπαθήσουμε να αναβαθμιστεί η συνεργασία μα μαζί του. Ε, θετικό μήνυμα αφορά κάποια έργα κοινού συμφέροντο όπω το πρωτόκολλο για τη συμμετοχή σε προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των υπηρεσιών, ακριβώ όπω και το κείμενο που εγκρίνουμε σήμερα, τεχνική συμφωνία, ωφελεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια όλα αυτά τα χαιρετίζουμε ιδιαίτερω. Ελπίζουμε δε ότι η συμφωνία θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την επικείμενη αποστολή τον Σεπτέμβριο στο Μπακού. Εδώ βάζω τελεία και αν έχετε τυχόν ερωτήσει, ευχαριστώ να απαντήσω. Ε, ευχαριστούμε, πρόεδρος. Για τη λεπτομερή αυτή παρουσίαση, κύριε Νικολάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ καταρχάς τους συναδέλφους Θέλω να ρωτήσω καταρχάς ποιος χρειάζεται το Αζερβαϊτζάν. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το Αζερβαϊτζάν όπως το Αζερβαϊτζάν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν και οι δύο πλευρές να βρουν τον τρόπο να βελτιώσουν την κατάσταση. Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω. Πριν από δύο χρόνια φαίνονταν μια παγωμένη σύραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν. Αλλά δεν χρειάζεται να αναζητούμε υπετίου και οι δύο έχουν ευθύνη. Ο Καύκασος και το Αζερβαϊτζάν έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικώς Χαίρομαι ιδιαίτερω που τώρα έχει ξαναρχίσει αυτή η διαδικασία για την ανοικοδόμηση τη εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν. Πριν από δύο εβδομάδε στον Πακού, ω μόνιμη αντιπρόσωπο, ε, επεσκέφθη και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Αλίεφ. Και είδα στο πρόσωπό του αποφασιστικότητα και βούληση για προσέγγιση και αποκατάσταση στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πολύ καλά μέσα στη διάθεσή μας για την ενοικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης ή τρέχουσες εξέλιξη περιλαμβανομένες και της κατάστασης σχετικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι νομίζω ευνοϊκέ και μπορούμε να συζητήσουμε ή τι άλλο έχουμε συνομιλητές. Για μένα η οικονομική κατάσταση δεν έχει τόση σημασία. Δεν αποτελεί, πιστεύω, κίνητρο για το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα η οποία τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και με βάση αυτά πρέπει να συνομιλούμε και όχι με βάση την οικονομική ευρωστία. Πρέπει να μιλούμε με αξίες και σε αυτό βλέπω μεγάλη βούληση από τους πολιτικούς, την κοινωνία των πολιτών, τον κοινό πολίτη. Γιατί είναι υπέρ της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. η παρουσία της είπα προσώπου Μογκερίνη επίσης ε, γέννησε πολλές προσδοκίες και γέννησε σεβασμό Είναι προς το συμφέρον μας πιστεύω να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να βρούμε έναν τρόπο να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτάν. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Μακάλιστερ, σκιώδηση ηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συμφωνούμε πιστεύω όλοι ο διάλογος οι συνομιλίες πρέπει να, να παραμένουν στο επίκεντρο των σχέσεων μας με το Αζερβαϊτζάν και θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε ευρωπαϊκές αξίες, κράτος δικαίου, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία. Πρώτον, όπως υπόθηκε ήδη, καλώς και εγώ, την απόφαση των αζερικών αρχών να αποφυλακίσουν επιτέλους ε, πολιτικούς κρατουμένους. Μήνυμα και σημάδι ότι η χώρα ε, πληρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις δυνάμει των Εθνών, των Εθνών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει και να κλεισμονούμε εκείνους που είναι ακόμα στη φυλακή και, τη σημασία, και να υπογραμμίζουμε πάντα τη σημασία του κράτους δικαίου και βέβαια την υποστήριξη των ε, οργανώσεων τι κοινωνίε των πολιτών στο Αζερβαϊτζάν. Ταυτόχρονα πρέπει το Αζερβαϊτζάν να συνεχίσει την ανάπτυξη αυτή τη στρατηγική συνεργασία και σε σχέση με την προμήθεια σε φυσικό αέριο. Τρίτον, ο Λεγόμενο τετραημερη πόλεμο πόλεμος 1η ω 4η Απριλίου του 2016 δείχνει πόσο ε, λεπτή και εύθραυστη είναι η κατάσταση στο, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε προσοχή λοιπόν στην κατάσταση αυτή πρέπει και προς την αρμενική όπως και προς την αζερική πλευρά να επισημάνουμε κάποια και να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Η αποφυγή της χρήσης βίας επίσης, ε, ο σεβασμός εδαφικής ακαιρεότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να επικαιροποιηθούν όπως υπόθηκε νωρίτερα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αζερβαϊτζάν, η συμφωνία εταιρική σχέση του 1979 ε, προσφέρει ακόμη ένα νομικό πλαίσιο, όπως είπαμε όμως χρειάζεται επικαιροποίηση για την εξεπερασμένη. Άρα θεωρώ ότι είναι καλό το ότι ανοίγουν και άλλοι διεύλοι επικοινωνία. Καλωσορίζω τις ε, πρωτοβουλίες της κυρίας Χάουταλα και του κυρίου Ντούλιτσα της Γεωργίας από το Euronest που επισκεφτήκαν τον Πακού για να ξαναρχίσει μια διακοινοβουλευτική συνεργασία ώστε το Αζερβαϊτζάν να επανέλθει στους σκόπους του Euronest και επίσης η Επιτροπή Βουλευτική με το Αζερβαϊτζάν για πρώτη φορά ύστερα από τέσσερα χρόνια θα συνεδριάσει τον Πακού εφέτος και το σημειώνω αυτό θετικά. Ευχαριστώ. Λόπες, ο έτερος συγητής και ο συγητής της Σοσιαλιστής Δημοκράτας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για μας αυτή παρουσίαση που μας κάνατε για την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Δεν είναι τυχαίο που αντιμετωπίζουμε το θέμα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερμπαϊτζάν μετά από τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασαν αυτές τις δυσκολίες τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνε οι δύο πλευρές για όλα αυτά. αλλά ήταν μια κάπω ιστερική απάντηση του Αζερμπαϊτζάν στι επικρίσει που διατύπωσε εναντίον του η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω ε, του Κοινοβουλίου σε ένα ψήφισμα που διατυπώσαμε και φυσικά και τη δική μας επιτροπή που ενέκρινε τα προγράμματα αυτά που τελικά ενέκριναμε. Η απάντηση της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν ήταν υπερβολική και τώρα πια υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον που εμείς το βλέπουμε θετικό να επανέλθουμε σε ομαλές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερμπαϊτζάν που να συνοδεύεται από βήματα προ τα εμπρό σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, απελευθέρωση ορισμένων πολιτικών κρατουμένων κτλ. Όπω όμω υπενθυμίστηκε, ακόμα πόρο απέχει η κατάσταση του Αζερμπαϊτζάν από το να είναι θετική. Υπάρχουν πολλοί ακόμα πολιτικοί κρατούμενοι, υπάρχουν πολλέ δυσκολίε σε ό,τι αφορά κράτο δικαίου, έκφραση ελεύθερη, ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι σοβαρά προβλήματα, γι' αυτό εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις που προωθούμε και πάλι με το Αζερβαϊτζάν για να συζητήσουμε για τα προβλήματα αυτά όπως έχει γίνει με την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν. Αναφέρθηκε στο παρελθόν ότι έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα και γνωρίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα πρόβλημα αυτοεκτίμηση στη συζήτησή μας, αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι πάντα έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε το ρόλο ενός παγκόσμιου παίκτη και να ασκούμε επιρροή και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει πραγματικά επιρροή πάνω στο Αζερβαϊτζάν. Είναι φανερό ότι υπάρχουν ε, συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή σταθερότητα. Αναφέρθηκε η σύγκρουση των τεσσάρων ημερών με την Αρμενία. Μας ενδιαφέρει ο διαπολιτισμικός διάλογος επίσης και μα ενδιαφέρει και η, στα, γεωστρατηγική πτυχή λόγω των πηγών ενέργειας του Αζερβαϊτζάν. Πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά εμείς ως παγκόσμιος εταίρος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την επιρροή μας. αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του Αζερβαϊτζάν έδειξε πως με κάποιες πιέσεις η Ευρώπη, και εδώ το Κοινοβούλιο μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα, μπλοκάροντας ορισμένα προγράμματα και εξηγώντα τη θέση μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ψήφισμα, μπορέσαμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα στο Αζερβαϊτζάν. Ακόμα βλέπουμε ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα εκεί, αλλά ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να στείλουν προς τη σωστή κατεύθυνση τη χώρα αυτή, που όπως εξηγήθηκε στην αρχική παρουσίαση, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της πτώσης του τιμή του πετρελαίου κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε μεγάλη εσωτερική πολιτική ασταθερότητα. Ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί μιλάμε σήμερα για το Αζερμπαϊτζάν. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα στα σταυροδρόμια διαφόρων συμφερόντων και το στρατηγικό ενδιαφέρον του για το Αζερβαϊτζάν θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον. Χρειαζόμαστε το Αζερβαϊτζάν και ως εταίρο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του και με ποιο τρόπο εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο και όχι όταν τα πράγματα πια έχουν εκφύγει κάθε ελέγχου. Χαίρομαι που τελικά έχουμε καταλήξει σε ένα επικοδομητικό διάλογο με το Αζερβαϊτζάν. Εγώ δεν ένιωθα καλά. Με την σκληρότητα που είχαμε δείξει στη σχέση μας. Με τη σκληρότητα αυτή δεν μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες αλλαγές στη στάση των εταίρων μας. Μόνο ο διάλογος και η ανεκτικότητα στο διάλογο επιτρέπουν να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Και εγώ θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την Κομισιόν και προς τον εισηγητή μας, όλους αυτούς οι οποίοι ανεπλάκησαν στην ανανέωση του διαλόγου μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια χώρα που υποστηρίζει τη δημοκρατία και το δυτικό κόσμο. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου εμείς δεν αντιπεριοδοποίησαμε το Αζερμπατζάν με τα ίδια κριτήρια όπως τις άλλες χώρες της περιοχής όπου υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό για την κοινωνία των πολιτών με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε πιο απότομη και σκληρή με το Αζερβαϊτζάν και ίσως και το Αζερβαϊτζάν έχει συμβάλει σε αυτή τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσπάθειά τους να δείξουν ότι είναι μια ισχυρή χώρα. Γιατί είχαν δημιουργήσει, έκαναν πολλές εκδηλώσεις, διοργάνωσαν μεγάλα γεγονότα, τα οποία τελικά μάλλον έπληξαν, παραβόητησαν την εικόνα του. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια προδραστική ε, λειτουργία στην ομάδα του Μίνσκ και σε σχέση με το πρόβλημα του Ναγκόνο Καριμπάχ το οποίο είναι ασυμμετρικό. Έχουμε μια χώρα τη οποία το έδαφο έχει τύχει κατοχή και εξακολουθεί να είναι υποκατοχή και έχουμε μια χώρα η οποία είναι η κατέχουσα. Για κάποιο λόγο και με λίγη φαντασία μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κράτος το οποίο έχει ασκεί την κατοχή αυτή είναι το, αυτό το οποίο εμεί ευνοούμε και αυτό οδηγεί σε κάποια προβλήματα. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα του Μίνσκ αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της Γαλλίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξαναπάρει πίσω αυτή την έδρα γιατί είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπω ότι ο πρόεδρος αρχίζει να κουράζεται, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. It's on purpose, but anyway, uh, thank you very much. Uh, Επίτηδες, αλλά εντάξει, κυρία Λόχπιλερ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και επίσης ευχαριστώ την υπηρεσία εξωτερική δράση για τις επιτυχίε της. Έχει βελτιώσει την κατάσταση για μερικού πολιτικού κρατουμένου αξιοσημείωτο. Και μάλιστα όχι σε σχέση με τους ε, πιο επιφανεί, αλλά και τους λιγότερο γνωστούς ακτιβιστές έχετε καταφέρει να εξασφαλίσετε την αποφυλάκησή τους. Όμως στην περίπτωση του Μότοφ, ο οποίος δικαιώθηκε έναντι των αρχών του Αζερβαϊτζάν, θα πρέπει με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπη, του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να αποφυλακιστεί. Τώρα λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβει εντατική δράση για την υπόθεση αυτή. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι θα ήταν καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Grand Prix στη Φόρμουλα 1 17 και 18 Ιουνίου για να πιέσετε να αποφυλακιστεί πριν από το Grand Prix. Και επίσης για τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και την ε, χρηματοδότησή τους. Δεν ξέρω αν ε, ε, μπορώ να το πω για όλους, αλλά εσείς έχετε στη θέση σας κάποια εκατομμύρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών μας λέτε. Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες λοιπόν. Ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ναι, και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε τις σημαντικές πρόοδους που σημειώθηκαν χάρη στις προσπάθειες της κυρίας Μογκερίνη, του κυρίου Λαμπρινίδη που εξασφάλισαν την αποφυλάκηση των πολιτικών ε, κρατουμένων στο Αζερπαϊτζάν Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλοι κρατούμενοι που ανέφερε και ο εκπρόσωπο τη υπηρεσία εξωτερική δράση και δεν μπορούμε να του ξεχάσουμε όπω ο Μαλδόλφη παραδείγματι αλλά και άλλοι. Γι' αυτό και το λόγο ψηφίζω, ψήφισα σήμερα αυτήν την έκθεση, γιατί νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά πρέπει και να επιμείνουμε να αποφυλακιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ε, ακόμη περισσότερο. Γιατί πρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο, πρέπει η κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσει το ρόλο που της ανήκει. Να υπάρχει λογοδοσία. Και εμείς να είμαστε παρόντες. Ρωτώ λοιπόν τον επρόσωπο της Επιτροπής. Τι ρόλο βλέπει η Επιτροπή να μπορεί να διαδραματίσει ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει τη δυνατότητα να καταπολεμήσει να αγωνιστεί κατά τη να αγωνιστεί υπέρ της λογοδοσίας, της διαφάνειας. Δεν είναι μόνο το θέμα των χορηγιών από τους χορηγούς, αλλά και ιδιαίτερη αποφυλάξη εκείνων των γενναίων που τόλμησαν να διατυπώσουν επικρίσεις και επιπλέον να ζητήσουν προδοσία. Είναι δύσκολο έργο. Δεν συμφωνώ με την προοπτική ότι έχει την ίδια υπετιότητα με το Αζερβαϊτζάν, όπως είπε η κυρία Νικολάη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν διστάζω βέβαια να επικρίνω την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν το αξίζει, αλλά προκειμένου δεν θεωρώ ότι αξίζει επικρίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ήταν υπεύθυνη για τη φυλάξη των ανθρώπων αυτών. Ούτε θα συμφωνήσω με τον κύριο Βάγκελ ότι ήμασταν πολύ σκληροί. Όχι. Αρχέ ακολουθούμε, αρχέ στηρούμε. Αυτό οφείλουμε να πράττουμε. Γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη που έχουν λοιπόν, εγκαταλείπουν τι αρχέ του. Και αρκετοί ε, ε, ε βουλευτέ και ευρωβουλευτέ. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώ εμεί πρέπει να δρούμε με αυτόν τον τρόπο. Να απαιτούμε δηλαδή αυτό που απαιτήσαμε. Και βεβαίως άλλαξε η κατάσταση χάρη σε αυτό, όπως υπογραφίστηκε. Και είδαμε και τα αποτελέσματα. Δεν αρκούν όμως. Και μπορεί να είμαι διτεθειμένη να δεχθώ ένα άλλο πλαίσιο σαν πειραματισμό για την ε, εξέλιξη και τις αλλαγές, αλλά δεν είμαι διτεθειμένη να υποχωρήσω σε σχέση με τις απαιτήσει που πρέπει να διατυπώσουμε στις αρχές του Αζερβαϊτζάν. μια ναι, κοινωνία πλούσια όπω το Αζερβαϊτζάν πρέπει να μπορεί να διαθέτει τους σπόρους τη ε, σε όλους και όχι μόνο σε μια κλεπτοκρατική ελίτ χωρίς λογοδοσία. Σας ευχαριστώ. Κιουτσίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σημαντική αυτή η χώρα από πολλές πλευρές. Και από την οικονομική πλευρά, ενεργειακή ασφάλεια και βέβαια όπω αναφέρεται και από πλευρά της ψηφιακής οικονομίας και για την πολιτική αεροπορία γιατί με επιτυχία άρχισαν να υλοποιούν τα διάφορα έργα με τις ε, γειτονικές χώρες, με τη Γεωργία, με την Τουρκία και επίσης έχουμε και στο Μέτσαμορ ε, το πυρηνικό εργοστάσιο και έχουμε πει και το πρόβλημα της Το και περισσότερο αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Για καιρό και περισσότερο ή αποτελεί έναν διάδρομο, έναν διάβλο για τα ενεργειακά. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται με την περιφέρεια αυτή, πώς θα αντιμετωπιστούν οι απειλές, πώς θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια, τέλος πάντων, το στεγανό αυτού του διαδρόμου. Ευχαριστώ. Κύριε Παντζέρη, για τον λόγο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Οφείλω να σας πω ότι ε, Έχω προβληματιστεί, έχω εκπλαγεί για αυτό που συζητάμε για το ε, Αφού ψηφίσαμε, συνήθως προηγείται συζήτηση της ψήφου. Πολύ συζητήσιμη αυτή η μεθοδολογία. Εγώ τώρα δεν θέλω να καταστρέψω το πνεύμα συνεργασίας που πρετανεύει στη σχέση με τη χώρα αυτή. Βεβαίω καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί πολιτικού ρεαλισμού ε, αυτό ε, κυβερνά ε, την στάση μας και ακόμα πάντως δεν έχω εμπιστοσύνη στην άργουσα τάξη της χώρας γιατί διαχρονικά έχουν δείξει ότι κάνουν πολλές κολοτούμπες και είπαμε ότι στην αρχή δημιουργούν ένα αλφα καλό όμως στη συνέχεια ακολουθούν άλλες λύσεις καταστολής. Φυσικά και δεν δίνουμε κανένα πράσινο φως, καμία επιταγή είναι λευκό, ε, τα προβλήματα σοβούν ακόμα στη χώρα. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα ανθρωπίνα δικαιώματα, θα πρέπει να αποφυλακιστούν ε, αυτοί που είναι ακόμα φυλακισμένοι και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα διευκολυνθεί η δράση των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει ο κύριος Έκλειστον να μας πει τι έγινε, τι έγινε επίσης ε, και με ε, το... Τι θα γίνει με τον Μπακού, εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1 και θα πρέπει να δούμε και να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει ότι εάν βάλουμε ως προϋπόθεση τις προϋποθέσεις η υλοποίηση αυτής της ε, έκθεσης θα πρέπει να τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις γιατί είδαμε κάποιο είδους ε, ανοιχτό πνεύμα αλλά δεν θα πρέπει ε, πέραν αυτού να ξεχνούμε τα προβλήματα τα οποία σου Ευχαριστούμε, λέει ο Κυρία Φωτίγκα. Και εγώ θα ήθελα, λέει η κυρία Φωτσίγκα, να ευχαριστήσω τον ομιλητή για την πλήρη αυτήν πληροφόρηση και να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη για την έκθεσή της που οδήγησε στην ψηφοφορία μας προηγουμένως στην ΑΦΕΤ. Σίγουρα χρειαζόμαστε το Αζερβαϊτζάν όπως και αυτή η χώρα μας χρειάζεται. Υπό έποψη ασφαλείας είναι μία από πολλές χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό έχει μια κοινωνία που είναι κοσμικού χαρακτήρα. Παρά όλες τις άλλες επικρίσεις που μπορούμε να διατυπώσουμε, θα πρέπει να δούμε τις θετικές χειρονομίες της κυβέρνησης του Αζερβαϊτζάν. Πρέπει τώρα να σκεφτούμε για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για επαφές, όχι μόνο διάλογο. Πιστεύω λοιπόν ότι παραμένουν πολλά πρακτικά θέματα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όχι σε απομόνωση, αλλά να τα εντάξουμε στην περιφερειακή συνεργασία. Πιστεύω όμως ότι και τα θέματα εσωτερικών και ο ρόλος ο σημαντικός της χώρας αυτής στο Νότιο Κάφκασο στο να ανασχέσει την κίνηση των ριζοσπαστών που πηγαίνουν στο Ισλαμικό κράτος είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ για το Αζερμπαϊτζάν, στην Επιτροπή Ασφάλειας και Αμήνας και νομίζω πρέπει να συνεχίσει το ενδιαφέρον μας για τη χώρα αυτή και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είδατε ήταν πολλά τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν από τους συναδέλφους. Ο κύριος Σόιμπλε λοιπόν θα μπορούσε να απαντήσει σε κάποια τουλάχιστον από αυτά τα ερωτήματα. Παρακαλώ. Thank, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολυπληθή σχόλια και τις ερωτήσεις. Φυσικά υπάρχει μια διαφορετικότητα στις εκτιμήσεις σας για το Αζερμπαϊτζάν. Ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλντερ για τη θετική αξιολόγηση της προσπάθειας της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που πράγματι πιστεύουμε ότι συνέβαλε στο να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά την κατάσταση των πολιτικών κατουμένων από την κοινωνία των πολιτών, την αντιπολίτευση και τους άλλους ακτιβιστές. Η πρόθεσή μας βέβαια είναι να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, όχι μονάχα να απελευθερωθεί ο Μαμάτοφ. Και άλλοι ακτιβιστές που δεν έχουν ακόμα απελευθερωθεί από τη φυλακή, θα θίξουμε το θέμα αυτό σε οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου αλλά και μεσαίου επίπεδου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε στο τέλος τα άτομα αυτά να απελευθερωθούν όσον ουπώ. Προσωπικά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Grand Prix της Φόρμουλα 1. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να έχουμε επιρροή σε ένα Grand Prix. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε μια ειδική ευκαιρία για να αναφέρουμε τα θέματα αυτά. Θα πρέπει εμείς να τα τονίσουμε σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως εν ώψη των διαπραγματεύσεων όταν αυτό θα πραγματοποιηθεί. Για την νομοθεσία για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Το αναφέραμε αυτό το θέμα σε μια προηγούμενη επαφή. Ο κ. Μέντιθ από την DGN το έθεσε με τον, στον κύριο Μαμαριάνοφ, τον αρμόδιο υπουργό σε αυτή τη συνάντηση και εμείς θα εξακολουθήσουμε γιατί αυτό θα προβλήματα στην χρηματοοικονομική μας υποστήριξη σε ορισμένες ΜΚΟ. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάπου 3 εκατομμύρια τα οποία δεν μπορούσαν να ε, εκταμιευτούν τώρα για σχέδια που έχουν να κάνουν με την κοινωνία των πολιτών. Λόγω αυτής της νομοθεσίας ελπίζω λοιπόν ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν θα βρουν έναν τρόπο για να τροποποιήσουν αυτή την νομοθεσία ώστε η δική μας υποστήριξη και των άλλων χορηγών προς τις ΜΚΟ να μπορέσει να διευκολυνθεί. Ο κύριος Λόπες τώρα, για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η κοινωνία των πολιτών θα μπορέσει να εξακολουθεί να αγωνίζεται κατά της διαφθοράς και να προωθεί το κράτος δικαίου, μόλις υπάρξει νέα συμφωνία θα εξυπηρετήσει αυτό το στόχο. Σε αυτή τη νέα συμφωνία θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το κράτο δικαίου και τη δημιουργία ισχυρά δημοκρατία στο Αζερβαϊτζάν. Μπορώ να σα πω ότι επίση εργαζόμαστε με τα μέλη της κοινωνίας, του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Συμμαχίας του Αζερβαϊτζάν. Έχουμε δώσει οικονομική βοήθεια σε πολλούς τομείς που έχουν να κάνουν με ακριβώς αυτό το θέμα, μία από τις προτεραιότητες. του ενιαίου πλαισίου συνεργασία, όπω το λέμε, είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα στο Αζερβαϊτζάν. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο εργαζόμαστε μαζί με του ομολόγου μα. Και το Αζερβαϊτζάν έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ την αδελφοποίηση. Υπήρξαν πολλά προγράμματα αδελφοποίησης πολλαίων με πόλεις στο Αζερμπαϊτζάν από το 2007, που είναι πολύ σημαντικό λόγω του επίπεδου συνεργασία μας. και χαίρεται το Αζερμπαϊτζάν για τη βοήθειά μας στα θέματα αυτά διδημοποίησης ή αδερφοποίησης. Ο κύριος Κιούτσουκ τώρα έθεσε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Ο νότιος διάβλος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι το πιο σημαντικό ε, εγχείρημα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, όπως ξέρετε, από τη στιγμή που ο διάβλος αυτός θα λειτουργεί, που ελπίζουμε θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, περίπου 10% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο μπορεί να καλυφθεί από το αέριο του Αζερβαϊτζάν. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο λοιπόν, αλλά περαιτέρω εμείς ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ για να προωθήσουμε το θέμα αυτό και υπάρχουν και οι προετοιμασίες των διαφόρων υποπρογραμμάτων που είναι εν και οι συναδελφοί μας από την TG Energy στην Κομισιόν εργάζονται εντατικά για το θέμα αυτό. Μπορώ να σας πω ότι τόσο κυρία Μογκερίνη όσο και ο αντιπρόεδρος της ο κ. Σεφτσοβιτ, ο οποίος είναι τα θέματα ενέργειας, ήταν παρόντες στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Νότιου Διάβλου στις 29 Φεβρουαρίου στο Μπακού και οι δύο τόνισαν ιδιαίτερα την σημαντική λειτουργία που έχει αυτό το project και τόνισαν τη σημασία των αζερμπαϊτζανικών αρχών. Αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Ο πολιτικός ρεαλισμός αναφέρθηκε από ένα Ιταλό συνάδελφο, δεν άκουσα καλά το όνομά σα. Νομίζω ότι είμαστε ρεαλιστέ όμω σε πολιτικό επίπεδο. Πολλά έχουν να γίνει, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προοπτικές για μια νέα συμφωνία που μπορούμε να επιτύχουμε όλα αυτά τα οποία μας είναι προσφύδει και αυτή η συμφωνία θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της μελλοντική μας συνεργασίας με το Αζερβαϊτζάν και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και την ανάπτυξη της δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τον μελλοντικό μας ρόλο και προφανώς θα μείνουμε σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως είπα στην εισαγωγή μου πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού για να κάνουμε σαφέστερα τα μηνύματά μας, γιατί τότε θα έχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εξωτερικές μας σχέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σούβαλ και όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή στη συζήτηση και προχωρώ τώρα στις ε, ε την ανταλλαγή απόψεων με την ΕΕΔ για την ομάδα εργασία για το εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Ο κύριο θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την Επιτροπή στην Ολομέλειά της για τη δουλειά μας. Τη δουλειά της Ομάδας Εργασίας από τη στιγμή που συστάθηκε με εντολή να εξετάσει τα θέματα των πέντε μέσων της εξωτερικής δράσης που θεσπίστηκαν με κανονισμούς και τακτική νομοθετική διαδικασία στις αρχές του 2014. Η εντολή της ομάδας μας έχει οικουμενικό χαρακτήρα, γεωγραφική φύση, θεματικά είναι ολιστική και εξετάζει δράσεις με βάση την αξία τους έως τα 132 δισεκατομμύρια για επτά Είχαμε 10 συνεδριάσεις πέρσι. Και η έκθεση που σας έχω διανύμει και γραπτός σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σας κουράσω για να διαβάσω κάθε λεπτομέρεια. Ξεκινώντας όμως θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα το προσωπικό της Επιτροπής για την υποστήριξη που προσέφεραν στη δουλειά μας. Η ομάδα μας προσπάθησε, επέτυχε και επιδιώκει πάντα να συνοψίζει τις εργασίες των συνεδριάσεων μας σε μια έκθεση που κατετέθη στον πρόεδρο Έλμαρ Μπροκ, ο οποίος επί τη βάση αυτών των εκθέσεων προβαίνει σε ανταλλαγή επιστολών με την αντιπρόεδρο Μογκερίνη ή τους επιτρόπους Πίμικα και Χάν ή σε άλλε περιπτώσεις μπορεί και να βρει ανταπόκριση από την Επιτροπή, δηλαδή να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα που έχει επισημάνει η ομάδα μας. Άρα δεν αποτελούσε αυτό σκοπό η σύσταση της, της ομάδας. Θελήσαμε να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Τα θέματα αφορούσαν εφαρμοστικές πράξεις, εγκάρσεις πολιτικές, Εξετάσαμε ζητήματα με συγκεκριμένη γεωγραφική εστίαση ευρωπαϊκή, στρατηγική παραδείγματι για το Ιράκ και τη Συρία, αντιμετώπιση του Ίσης, ε, την Ισία, Παλαιστίνη, Βιρμανία, Μιανμάρ. Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα από τη δουλειά μας και σημαντικό θα ήταν, πιστεύω, να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τον πολύ θετικό τρόπο με τον οποίο υποστήριξαν τη δουλειά μας και την ενημέρωση που μας βοήθησε να καταλήξουμε σε εις βάθος συζητήσεις. Ένα θέμα δεν έχω περιλάβει γραπτός στην έκθεση, αλλά θα την κλειτώσετε, θα σας το πω. Το συμπέρασμά μου είναι πως δεν είναι ικανοποιητική η παρούσα μορφή και σύσταση της ομάδας εργασίας. Άρα, σας δίνουμε βέβαια την ευκαιρία για να δείτε την επισκόπηση των εργασιών, αλλά για μένα το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το πείραμα στο οποίο συμφώνησε αυτή η ομάδα εργασία με τη, κατά τη σύστασή δεν απεδείχθη απολύτως επιτυχε. Θα θυμάστε πιο πριν είχαμε διάφορες και συγκεκριμένε ομάδες εργασίας που εξέτασαν η κάθε μία ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Οι οποίε de facto είχαν δημιουργήσει ομάδες σκληρού πυρήνα μικρές, μικρότερες ομάδες, 3-4-5 βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες που εργάζονταν εντατικά ε, πάνω σε καθένα από αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Η ομάδα εργασίας υποτίθεται ότι θα εξετάζει ταυτόχρονα όλα αυτά τα μέσα. Και δεν μπόρεσε να το πράξει κατά τρόπο που για μένα θα θεωρούνταν ικανοποιητικός. Και λόγω του εύρους του πεδίου εργασιών και της φύσεως, αλλά και γιατί ήταν μάλλον χαμηλή η προσέλευση και παρουσία των συναδέλφων κατά μέσο όρο. Τρία μέλη της ομάδας εργασίας, πέραν των εκπρόσωπο του, του εκπροσώπου του Προέδρου, του Προέδρου θα έλεγα, και εγώ προσπάθησα να είμαι πάντα παρόν, αλλά πέραν αυτού τρεις συνάδελφοι μπορούσαν να είναι παρόντες στο ίμιση των συνεδριάσεων. Ε, αυτό δεν είναι δουλειά. Δηλαδή. Θέλω να το πω αυτό ξεκάθαρα, να λέω ότι δεν είχε κανένα νόημα η δουλειά μα. Μπορέσαμε να φέρουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν ήταν παραγωγική δουλειά μα όπω το θέλαμε. Εάν θέλουμε να έχουμε μια επισκόπηση και επιτήρηση, υποπτία κοινοβουλευτική, πρέπει να αναλάβει αυτό το έργο ήδη η Επιτροπή και όχι η Ομάδα Εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εύστοχε οι, παρα... οι παρατηρήσει σα, η κυρία Λόζιν και η κυρία Λόχ Μπίλτερ, γιατί και οι δυο σα έχετε συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα. Λόζιν, σα ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με πάρα πολλά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπιτικόφερ προηγουμένως. Θα ήθελα Καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μπιτικόφερ, όπως και την αρμόδια γραμματεία της ομάδας αυτής εργασίας και για την προετοιμασία των συνεδριάσεων αυτής της ομάδας εργασίας. Ως είδαμε, ιδίως με τα έγγραφα τα οποία μας παρουσίασε ο κύριος Μπούτι Κόφερ, Υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα του θέματος αυτού, το οποίο μας απασχολεί και το, η ομάδα αυτή εργασίας θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου. Έχω λάβει μέρος στο, στην ομάδα εργασία για το μέσο σταθερότητα και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να εργάζεται κανεί σε ένα τόσο διαφοροποιημένο πλαίσιο. Αλλά έχει επιτευχθεί χάρη στην εργασία της γραμματείας και την ηγετική ικανότητα του κυρίου Μπουτικόφερ να κάνω κάποιες διαδικασίες διαφανέστερες. Παρά όλα αυτά όμως, πρέπει να πω ότι η οργάνωση και η προσπάθεια που έγιναν σε αυτή την ομάδα εργασία δεν εστέφθησαν υπό πραγματικής επιτυχίας ακριβώς γιατί πολλοί από τους βουλευτέ δεν έχουν λάβει μέρο και δεν έχουν συμμετάσχει στο βαθμό του επαρκού. Γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία χρειάζονται παρουσία των βουλευτών. Έχουμε λοιπόν την απόψη η οποία αναφέρθηκε τότε όταν γινόταν διαπραγμάτευση στο μέσο σταθερότητας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα ελέγχου και να υπάρχει η διαδικασία συναπόφασης και όχι απλώς διαβούλευσης όπως κάνει, παραγωγός χάρη, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για τα θέματα προϋπολογισμού. Ξέρω ότι αυτό θα σήμαινε σημαντικό άχθος, σημαντική προσπάθεια και εργασία για να πραγματοποιηθεί, όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη <coughs> την κατάσταση που επικρατεί και τα κονδύλια, το ύψος των κονδυλίων που βρίσκονται σε αυτό το εργαλείο, την πολυσχηδή και πολύπλοκη σφαίρα εφαρμογής αυτού του Μέσω την έλλειψη επαρκούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών της Κομισιόν θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία αυτού του ε, μέσου που ο έλεγχος του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλήρως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λόχμπιλντερ. Είμαι σύντομη γιατί δεν έχω πολλά να προσθέσω στην έκθεση του κυρίου Μπούτικοβερ. Και η Επιτροπή μου μου είπε να τονίσουμε στο περιεχόμενο το θέμα της, του κοινωνικού των δικαιωμάτων επίσης. Το θέμα είναι το ότι θα πρέπει να δούμε την υπόθεση της συμμετοχής των βουλευτών, γιατί είχαμε μόνο την ομάδα εργασίας στην τελευταία θητεία και εγώ θα προτιμούσα εάν έχουμε αλλαγές να επιστρέψουμε στην ε, άλλη μορφή οργάνωσης γιατί θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες επεξεργασίας όλων των χρηματοδοτικών μέσων. Άρα θα πρέπει ε, με τον Πρόεδρο, με το Δημιουργικό Προεδρείο, να δούμε σύντομα το θέμα. Και έχουμε και άλλη μια αυτή που ασχολείται με τον ΟΗΕ. Μόνο μία συνεδρίαση έγινε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος και να οργανώσουμε κάποιες συναντήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Και κατόπιν τα αποτελέσματα, όπως έγινε και με τον ΟΗΕ, να περάσουν στις γνωμοδοτήσεις στη ΣΑΦΕ. Το πρώτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε, λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και πρόκειται να τις διαβιβάσουμε αρμαδίως και θα συζητηθούν τα όσα είπατε στο διευρυμένο Προεδρείο. Αλλά και στην Επιτροπή βέβαια. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Το τελευταίο σημείο είναι η αναφορά των τρίτων χρόνων των οποίων ε, οι πολίτες θα πρέπει να κατέχουν θέση διαβατηρή όταν ε, περνούν τα εξωτερικά σύνορα και επίσης τις χώρες ε, των οποίων οι πολίτες απαλλάσσονται αυτής της ε, υποχρέωσης. Συγκεκριμένα θα συζητήσουμε για το Κόσοβο. Ο κύριος Σόλτες αντί για την κυρία Λούνατσεκ. Θα έρθει σε λίγο κύριος Σόλτες. Μόλις 7 η ώρα θα αρχίσει το μάτσα απόψε. Πρέπει να σας ενημερώσω. Exactly. Ah, Ό,τι θέλουμε μπορούμε να ζούμε. We have some colleagues here who have asked for the floor. συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Και μέχρι να έρθει ο κύριος Σόλτες, ε, ζητώ από τον κύριο Άνταξον να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Σουηδία, από όπου προέρχομαι, Εμείς που υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα προσθέμενες αξίες για να πείσουμε τους συμπολίτε μας για την ανάγκη να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυθυρημένοι αριθμοί, οι γενικέ δηλώσεις δεν επαρκούν. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο οι πολίτες μας μπορούν να το κατανοήσουν, να συνδέονται με αυτά οι καθημερινές ζωές τους. Σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για το λαό του Κωσυφοπεδίου. Όλοι οι γείτονές τους στα Βαλκάνια έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν με δίχως βίζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Κομισιόν. Ο, ε, επειδή η Κομισιόν θεώρησε ότι τα προαπαιτούμενα έχουν επιτευχθεί. Στην περίπτωση όμως των Κωσοβάρων όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να είναι πάντα ειλικρινή σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέλλον του Κωσοφοπέδιου. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα μόνο αν εγκριθεί η φιλελευθερωποίηση στις ε, προξενικές θεωρήσεις. Η Συμφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας προβλέπει και την ενίσχυση των ευκαιριών εργασίας, υποστήριξη των ε, μεταρρυθμιστό στροφών δυνάμεων στο κοσφοπέδιο και δίνει τη δυνατότητα να γίνουν αυστηρά μέτρα για να μπορέσουν να προσποριστούν οι πολίτες του κοσυφοπεδίου ε, θετικά στοιχεία. Χαιρετίζω λοιπόν όλα αυτά. Χαιρετίζουν όλα αυτά μάλλον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατανοεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας μηχανισμός εποπτείας στην εποχή μετά από τη φιλελευθεροποίηση και τη δυνατότητα να υπάρξουν ad hoc ενέργειες. Τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να εμποδιστεί η παράνομη μετανάστευση. Και επίσης καταγράφουμε τις υποχρεώσεις του Κωσυφοπεδίου σε σχέση με την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και τον αγώνα κατά του εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Το ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, έχει κατ' επανάληψη αναφέρει ότι εμείς θα βασιστούμε στην αξιολόγηση της Κομισιόν και με μεγάλη χαρά θα υποστηρίξουμε την άρση της υποχρέωσης για προξενική θεώρηση για τους πολίτες του Κωσόβου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άντακ Σόν. Ο κύριος Σόλτες έχει έρθει, οπότε μπορώ να του ζητήσω να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα πρώτα για άλλη μια φορά να σας αναφέρω ότι δυστυχώς η Ουλρίκη δεν μπόρεσε να έρθει διότι είχε μια σοβαρή εγχείρηση η μητέρα της, οπότε και εγώ θα την αντικαταστήσω. Οπότε όσον αφορά αυτή την κατάργηση της βίζας για το κοσυφοπαίδιο, θεωρούμε θετική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να ισχύσει αυτό το μέτρο για τους Κωσοβάρους. Και επίση θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο που θέλουμε επίση να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτή η διαδικασία και να τεθεί ο τροποποιηθής κανονισμός σε ισχύ ούτως ώστε ο κόσμος να ωφεληθεί. Κατάρριξη της είναι πάντως ένας τρόπος ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη επαφή των ανθρώπων και έτσι θα έρθει η χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια. Από το 2010 που οι πολίτες της αντίθετα με τους πολίτες των άλλων χωρών δεν, μπορούν, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Οπότε θα πρέπει να πάρουν βίζα για να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι είναι πολίτες δεύτερη κατηγορίας. Άρα παρακαλούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να πληρούν τις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση δεν θα καταπολεμήσει διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα. Η δε αντιπολίτευση θα πρέπει να επιψηφίσει την, συνθ... την κύρωση της συνθήκης ε, για τα σύνορα της συνθήκης με το Μαυρό Βούνιο. Πρέπει να εγκρίνουμε το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση μέσω της κυρίως Αρμόδιας Επιτροπής και Συμβούλιο και Επιτροπή να ολοκληρώσουν την έγκριση μια που οι προϋποθέσεις θα πληρούνται. Έχει κάνει μεταρρυθμίσεις η χώρα. Έχει προοδεύσει κατά το 2014 και πληρεί το 95% των προϋποθέσεων που έχουν εταχθεί για το χάρτη πορείας που αφορά τη Βίζα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάθε χώρα. Όπως ισχύει τώρα για Κοσκοπέδιο, για Γεωργία, για Ουκρανία και για Τουρκία, θα πρέπει να δικαιούται την ε, κατάραξη της θεώρησης αλλά κάθε περίπτωση να κάνετε χωριστά. Και όχι όλοι μαζί σαν πακέτο. Και τώρα, ο κύριος Παντζέρη δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω. Πάντως σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να τα με την καινούργια υπεύθυνη της αντιπροσωπείας της Ένωσης εκεί ή στην Πρίστινα. Νομίζω ότι έχει πάρει καλό δρόμο η υπόθεση αυτού του μέτρου. Μια που είπαμε επανειλημμένα ότι θέλουμε να πλησιάσει περισσότερο στην Ένωση η χώρα. Υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν πέραν των ε, προϋποθέσεων που ακόμα δεν πληρούνται από τις αρχές της χώρας. Άρα χρειάζεται και μια αποφασιστική πολιτική μεταρρυθμίσεων τόσο ώστε η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει με τις σχετικές προσπάθειες και να ολοκληρώσει την προσέγγιση και σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει νόημα αυτό το μέτρο, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει οι αρχές χώρες να καταλάβουν τι γίνεται και να προχωρήσουν προς την, προς την ε, τήρηση αυτών των προϋποθέσεων. Και ο Τζαμπάσκη τώρα ζητώ λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόσκο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλωσορίζω το πνεύμα των ε, τοποθετήσεων των σε σχέση με την απελευθέρωση και υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίου. Έχω δώσω κάποιε ανησυχίε. Ίσως η Επιτροπή σπέβδει, υπερβολικά ε, να λάβει αυτέ τι αποφάσεις. Στην έκθεσή μα για το κοσφοπέδιο είχαμε σημειώσει πριν από ένα χρόνο ότι δεν είχε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις σε σχέση με τη συμφωνία με το Μαυροβούνιο, το Κοσφοπέδιο. Και αυτό είχε να κάνει και με το... Η διαδιπίστωση ίσχυε και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι λοιπόν και της διαφθορά. Έτσι λοιπόν το Κοσφοπέδιο πλέον έχει πάρει φήμη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται ακραίοι του Ισλαμικού κράτους παραμένουμε αμέτωχοι θεατές, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία δράση. Χώρες οι οποίες δεν κινδυνεύουν ε, από πόλεμο βλέπουν να καταφτάνουν σε αυτές μαχητές από το κοσφοπέδιο. Γι' αυτό διαφοροποιούν μεταξύ μεταναστών προσφύγων, παράτυπων μεταναστών η Γερμανία, η Αυστρία και γι' αυτό αρνούνται την είσοδο σε επικόστικο του Γιατί Γιατί προσπαθούν να καταπολεμήσουν τους από αυτούς μαχητές. Αποτελέσματα όμως από ό,τι λένε και τα Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πληροφορίες για 500 που έρχονται προς την Ευρώπη για να σχηματίσουν τάγμα του ΙΚΙΛ. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση πολύ σοβαρή, μια κατάσταση πολύ ανησυχητική. σε σχέση και με την ε, Γεωργία και την Ουκρανία, για τις οποίες εγώ υποστηρίζω την ε, απολευθέρωση υποχρέωση θεώρησης και θα, θα απόσχω. Ευχαριστώ κύριο Σπίτσουλα, ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας που καλύπτει και το κοσφοπέδιο, παρακαλώ. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με το κοσφοπέδιο σχετικό με την απελευθέρωση ε, της θεώρησης τον Ιανουάριο του 2012 και προσδόρισε την ίδια χρονιά ένα φιλοπορία στι προποθέσει που θα έπρεπε πριν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση του κοσφοπέδιο να εκπληρώσει και ταυτόχρονα ε, ήρε την ε, σε σχέση με τη θεώρηση, λέγοντας μεν ότι, ε, ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κοσφοπέδιου, αλλά ορίζοντας προϋποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής. Τη στιγμή όπου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα καταθέσουν τις προτάσεις του, το κοσφοπέδιο θα πρέπει να έχει κυρώσει συμφωνία διευθέτησης με το Μαυροβούνιο. Δεύτερον, θα έχει θα πρέπει να έχει προχωρήσει κατά καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται λοιπόν για τεράστια ε, ενθάρρυνση πιστεύω προς το κοσφοπέδιο να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του και την πρόοδο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σημειώνω πάντως ξεκάθαρα ότι τη σύσταση για την απαλλαγή την αξίζει το κοσφοπέδιο. 90 προϋποθέσεις έχει εκπληρώσει 40 περισσότερες από τα λοιπά κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. και δεν ε, φαντάζομαι να προκύψει πρόβλημα λόγω εσωτερικών εντάσεων και σχέσεων με το Μαυροβούνιο. Σε σχέση με την επίσημη πολιτική ορισμένων κατορμαλών που δεν θέλουν να γνωρίσουν το Μαυροβούνιο, το Κοσμοπέδιο, ελπίζω αυτό να μην ε, μας οδηγήσει σε οψοδρομήσεις. Υπάρχουν πολλά μελήματα ιστορικής πολιτικής στην περίπτωση αυτή προβλήματα που δείχνουν και μία επικοδομητική στάση από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει η δυναμική που έχει καθιδρυθεί στη χώρα. Η χώρα της Ευρώπης που έχει τον πιο νεανικό πληθυσμό δεν πρέπει να μείνει το χαμένο κομμάτι του μοσαϊκού. Το Κωσφοπέδιο είναι η μόνη χώρα μεταξύ πόντου και ατλαντικού, τις οποίες οι κάτοικοι δεν μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Σουίτσα, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ο κύριος Πίτσουλα, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας, είπε πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Και είναι αυτά που είπε και ο πρόεδρος μας. Εμείς πρόσφατα είμαστε στο Κωσυφοπαίδιο, έχουμε παρουσιάσει μια έκθεση στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και τα εμπόδια αυτά πραγματικά υπάρχουν και μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε στην εξαίρεση από προξενικές θεωρήσεις. Και το έχουμε τονίσει και προς τους ομολόγους μας κοινοβουλευτικούς και τα άλλα Ινστιτούτα του Κόσοβο. Ξέρουμε πόσα είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Κόσοβο και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο και ξέρουμε ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έχουν εδώ και πολύ καιρό πάψει να συνεργάζονται ακριβώς εκεί που είχαν αρχίσει και πάλι το έργο της και χάσαν ευκαιρία λοιπόν να συνεργάζονται. Νομίζω πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και καθεστώς των Δήμων που να αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία. Πρέπει να καταλάβουν οι αρχές του Κόσοβου ότι αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, ακόμα και αν ήταν ένα κριτήριο το οποίο δεν εφαρμόστηκε στις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσα στα πλαίσια της φιλελευθεροποίησης του που ξενικό θεωρήσεων. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στο Κόσοβο να μπορέσουν να πάρουν στα σοβαρά τα εγχείρηματα που πρέπει ακόμα να φέρουν σε πέρα πλαίσια της διαδικασίας για τη φιλελευθερωποίηση των ε, προξενικών θεωρήσεων και στην σύνολη διαδικασία προσχώρησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρώτο, Η κυρία Γκαμπριέλα Σμιτ, η οποία είναι αρμόδια για την ε, Βελαρούς, Μολδοβία, Ρώσια, Ρωσία, Ουκρανία και Κάμπο Βέρντε σε ό,τι αφορά την πολιτική προξενικών θεωρήσεων. Και το 25 φυσικά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με ακούτε και τον συγητή για τη θετική του άποψη και για την υποστήριξη της πρότασης Κομισιόν. Φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται ακόμα να εκπληρωθούν δύο benchmarks και είναι δύσκολο να μπορέσουν να εκπληρωθούν άμεσα από το κοσφοπέδιο Ελπίζουμε όμως ότι τα προβλήματα με την αντιπολίτευση μπορούν να ξεπεραστούν. Ξέρουμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ξέρουμε ότι το κοσφοπέδιο εκπληρεί 93 από τα 95 benchmarks ή τα τελευταία λοιπόν βήματα τα οποία εκκρεμούν και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να περάσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ την υποστήριξή σας, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Κύριε Κουκ, Καν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να σα εκπίξω γιατί σήμερα το πρωί συζητήσαμε και εξαντλήσαμε το του Κόσμου Πεδίου τότε που μιλούσαμε με την επικεφαλής της Αντιπροσωπής Ένωσης. Απλώς ε, σε συνέχεια το με κυρία Σουίτσα. Θέλω να σα πω ότι η Κόσοβάρη ε, παραπονιούνται επί πολύ καιρό ότι βρίσκεται σε μια νησίδα στα Δυτικά Βαλκανία, ότι είναι απομονωμένη, ότι φύστανται διακρίσεις σε σχέση με τους άλλους που μένουν ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και ε, δίκιο, αλλά το θέμα είναι ότι όταν θεσπιστεί η κατάργηση τις ε, βίζες, τότε θα πρέπει να λύσουν και ζητήματα και το ξέρουν. Εγώ συμφωνώ με την κατάργηση της βίζας. Όταν και αν λυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν τι πρέπει να πετύχουν. Ε, τότε θα συμφωνήσουμε την κατάργηση και στη τα διαβατήρια. Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζω ότι η προθυμία και τροπολογίες είναι 21η Ιουνίου το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ στις 7 Ιουλίου. Σε έκρηκτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Και η ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει στις 12 Ιουλίου. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 27 Ιουνίου ενεστώντας τους και σας ευχαριστώ. Πέρα στις συνεδρίες Thank you very much. Now we can go and watch the, the... Ε, τώρα μπορούμε να πάμε να δούμε το ματσάκι. yes. Austria versus Hungary, not Austro-Hungary against somebody else, as Otto von Habsburg has asked.